colleagues. Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ καθίστε, κύριε και κύριοι. Επιτρέψτε μου να σας ε, παρουσιάσω το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι η ανταλλαγή απόψεων με τρεις εξέχοντες προσκεκλημένους μας, οι οποίοι εκπροσωπούν τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα μας είναι η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Διεθνού Στρατηγικής στα πλαίσια της ασφάλειας και άμυνας. Θα ξεκινήσουμε με τη γενική παρουσίαση της ε, διεθνούς αυτής στρατηγικής, της σφαιρικής στρατηγικής και εδώ ο κύριος Μόλιναρ που είναι, εκτελείται καθήκοντα διευθυντή, Μετάρχη μάλλον, της CMPD DAE στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχείριση κρίσεων δηλαδή και σχεδιασμός. Επίσης έχουμε το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης, τον Υπογενικό Διευθυντή, το Γενικό μάλλον Υποδιευθυντή της DigiGrow, τον κύριο Πιέρ Ντελσό. Και τελευταίος αλλά όχι λιγότερος σημαντικός, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ο κύριος Μούιρα. Με συγχωρείτε για την προφορά σας, είναι πολύ δύσκολο να προφερθεί σωστά, είναι σκοτσέζικο το όνομα. Δύσκολη προφορά. Ε, πώς θα διαρθρώσουμε τη συζήτηση. Πρώτα, παρουσιάσεις από, από τον εκπρόσωπο της ΑΕΔ για την όλη έννοια της σφαιρικής διεθνούς αυτής στρατηγικής. Έπειτα ο κύριος Ντελσό, ο Γενικός Ποδιευθυντής και μετά ο κύριος Μουρ θα παρουσιάσουν την ε, φάση της υλοποίησης. Όπως ξέρετε από τον Ιούλιο φέτος η κυρία Μογκερίνη παρουσίασε την σφαιρική, τη διεθνή στατηγική. Τώρα έχουμε περάσει στη φάση της κατάρτισης προγραμμάτων δράσης. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με μια γενική παρουσίαση και μετά θα περάσουμε στην φάση της προετοιμασίας για να δούμε πώς θα γίνει και η υλοποίηση. Κύριε Μόλιναρ, ευχαριστώ πάρα πολύ να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα επικεντρωθώ στις παραμέτρους άμυνας και ασφάλειας της διεθνούς στρατηγικής, η οποία αφορά, η οποία αφορά διάφορες εργασιακές ε, κατευθύνσεις, ε, όπως ε, η ανθεκτικότητα του συστήματος άμυνας που θα έχουμε. Και εδώ θα επικεντρωθώ σε ορισμένες μόνο ο στόχος της γενικής, της τη εκπροσώπου είναι να υπάρξει ένα πρόγραμμα υλοποίησης για την άμυνα και την ασφάλεια που θα αποτιμήσει τον αντίκτυπο της σφαιρικής στρατηγικής σε αυτές τις δύο παραμέτρους. Η δουλειά αυτή γίνεται παράλληλα με άλλες, ε, άλλους τομείς εργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια. Το πρόγραμμα δράσης για την άμυνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μία, για το οποίο θα μιλήσουν και οι συνάδελφοι βεβαίω. και υπάρχει και η δουλειά που γίνεται για την υλοποίηση της κοινή δήλωσης ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ που υπογράφηκε στη Βαρσοβία. Αυτά είναι τα στοιχεία του προγράμματος, σε τρεις πυλώνες που θα οργανώσουν την εργασία μας αυτό το εξάμενο και για, το, για τους οποίους θέλουμε αποτελέσματα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν τη δουλειά μας για αυτό το πρόγραμμα εφαρμογής και υλοποίησης, το οποίο χοντρικά θα έχει δύο βασικά τμήματα. Με ένα ανώτερο επίπεδο φιλοδοξιών για την ε, κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, όπως προκύπτουν από τη σφαιρική στρατηγική και ε, τους νέους στόχους, τα αποτελέσματα για να φτάσουμε σε αυτό το ύψος φιλοδοξιών και στην πράξη. Έχουμε σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και περιμένουμε τις αποκρίσεις τους. Στόχος της είπα της εκπροσώπου είναι να παρουσιάσει το πρόγραμμα υλοποίησης στους υπουργούς τον Νοέμβριο στις 14 και 15 Νοεμβρίου στο Συμβούλιο. Νέο επίπεδο φιλοδοξιών λοιπόν. Αυτό θα είναι η θεμέλια λήθος για το πρόγραμμα υλοποίησης, το οποίο θα διοργανωθεί γύρω από τρεις στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες εκπηγάζουν από τη σφαιρική στρατηγική. Πρώτον, βελτίωση της δυνατότητας απόκρισης σε κρίσεις και συγκρούσεις. Δεύτερον, ενίσχυση Τη ε, δυνατότητας, της ικανότητας μάλλον, να ε, συμβάλλουμε στην οικοδόμηση δυνατοτήτων στα κράτη που έχουν πληγεί από κρίσεις και το τρίτον, προστασία της Ευρώπης. Αυτό μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι η προ... καινούργια, η νέα εξέλιξη μεταξύ των τριών προτεραιοτήτων. Εδώ δεν μιλάμε για συλλογική άμυνα, κοινή άμυνα ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι που το έχει αναλάβει ως όλο το ΝΑΤΟ για τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτό, για τους συμμάχους δηλαδή. Θέλουμε συνεργασία, σχέση συνεργασίας με εσωτερικούς φορείς σε έναν άξονα παρακολούθηση τη εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια ταυτόχρονα. Για τι απειλέ, στον κυβερνοχώρο, στη θαλάσσια ασφάλεια, στα σύνορά μα και ίσω και στο άρθρο 42.7, την αμοιβαία συνδρομή και τη σχετική ρήτρα. Το σημαντικό που θέλω να πω εδώ είναι ότι έχουμε μεν τρει προτεραιότητε, αλλά δεν αλληλοαποκλείονται. Οι εξωτερικέ παρεμβάσει και επιχειρήσεις μπορεί να έχουν απότερο σκοπό να τονώσουν και να ενισχύσουν την ασφάλεια στην, την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη. Μιλάμε για επιχειρήσει στη Μεσόγειο ή εμέσως αντιμετωπίζοντα άλλε ασταθεί περιοχέ στην ευρύτερη γειτονία μα. Να τονίσω επίση, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι μιλάμε και για στρατιωτικό και για πολιτικό επίπεδο φιλοδοξιών, σε επίπεδο στρατού και πολιτών δηλαδή. Καλύπτεται και η πολιτική διάσταση τη κοινή πολιτική ασφαλεία και άμυνα με επιχειρήσει που αφορούν του πολίτε πολλέ φορέ. Συνεργασία με εταίρου, ε, αναπόσπαστο τμήμα αυτή τη δουλειά. Από τη μια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει περισσότερε ευθύνε ε, στην αξιολόγηση αυτών των ζητημάτων. Από την άλλη, όμω, πρέπει να βοηθά και το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ στις δικέ του δυνατότητε απόκριση. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αντιφατική σχέση. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για δράση, διαφορετικά στοιχεία εδώ, ένα, προτεραιότητες ω προ τις δυνατότητές μας, οι οποίες θα εξαρτηθούν από αυτό το επίπεδο φιλοδοξών που έχουμε ορίσει, Αυτά όλα περιλαμβάνονται ήδη στην ε, ανάλυση της ε, σφαιρικής στατικικής και θα πρέπει να επικοινωθούν και τα κράτη-μέλη. Μετά, η δουλειά για την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας, αυτό νομίζω είναι δουλειά και, της, ε, και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του ΕΝΤΑ, και επίσης υποδομές και εργαλεία για να μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο φιλοδοξιών που έχουμε ορίσει. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμογής και υλοποίησης παραπομπές γίνονται εδώ στην δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Έχουμε παραπομπές στα, στις μονάδες, στα, τις μάχημες μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συλλογική στατικική απόκριση σε απειλές για την Ένωση. Και φτάνουμε και στη δέκατη επέτειο τώρα αυτών των ε, μάχημων μονάδων, οι οποίες έχουν αρχίσει ε, πλήρως να λειτουργούν από το 2007. Αλλά πρέπει να αποσταλούν και σε κάποιες πραγματικές επιχειρήσεις ακόμα. Ε, εντείνονται προσπάθειες και θα το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη πώς μπορούμε να το προωθήσουμε. Χρηματοδότηση και άλλο σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να υπάρξει απαραίτητη χρηματοδότηση, κάλυψη για να πετύχουμε το επίπεδο φιλοδοξιών μας και να είμαστε αξιόπιστοι. χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, με του σχετικού μηχανισμού και τα εργαλεία που γενικότερα έχουμε στη διάθεσή μα. Τέλο, αναφορέ έχουν γίνει στη μόνιμη δομή συνεργασία μας διάταξη τη συνθήκη που μπορεί να επιτρέψει να αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξιών και δεσμεύσεων των κρατών μελών. Όμω, από την οπτική γωνία των υπηρεσιών μα, εξαρτώμεθα πραγματικά από τα ίδια τα κρατη Εκεί να πρέπει να έρθουν με πρωτοβουλίε σε εμά και με προτάσει για προγράμματα. Είναι μια διαδικασία που θα την κινήσουν τα κρατη τα ίδια. Αλλά θέλουμε να διερευνήσουμε όλε τι δυνατότητε που έχουμε μπροστά μα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματο εφαρμογή και υλοποίηση. Και πάλι ο γενικό στόχο είναι να έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε τον Νοέμβριο στους υπουργού στο Συμβούλιο Άμυνας και βεβαίως και το Δεκέμβριο για τη Σύνοδο. Τότε περιμένουμε να έχουμε άλλα σημαντικά αποτελέσματα για να παρουσιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σταματήσω εδώ. Thank you, sir. Ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στη φάση της υλοποίηση. Με ερωταπαντήσεις και για τα δύο θέματα, ώστε πρώτα να έχουμε μια συνοπτική εικόνα της σφαιρικής στρατηγικής και της υλοποίησής της. Για αυτό το λόγο θα δώσω το λόγο στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Grow, τον κύριο Πιερντελσό. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Όταν μιλάμε για άμυνα είναι σημαντικό να μιλάμε σε, με όλους τους ε, ε, πρωταγωνιστές και το Κοινοβούλιο είναι ένα από τους πρωταγωνιστές πριν περάσουμε στη φάση εκτέλεσης. Ε, όπως ε, σας είπε και ο συναλφός μου, ε, έχουμε τρεις άξονες, την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, το Ευρωπαϊκό Δράσης, Πρόγραμμα Δράσης Άμυνας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τώρα γιατί εργαζόμαστε στο Πρόγραμμα Δράσης. Γιατί αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ικανότητες στην Ευρώπη και στο μέλλον, χρειαζόμαστε μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Και γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία περνάει δύσκολες στιγμές για διάφορους λόγους. Δεν θα επεκταθώ, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε την αμυντική βιομηχανία, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε τις ικανότητες, στρατικές ικανότητες που θα χρειάζονται τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους. Οπότε εργαζόμαστε επί αυτού του σχεδίου δράσης ε, ε, για την άμυνα που θα υιοθετηθεί στις 30 Νοεμβρίου, σε μερικές εβδομάδες. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Άμυνα δεν είναι αυτός σκοπός. Ε, θα απαριθμεί μια σειρά δράσεων οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν στο μέλλον. Και σε αυτό το σημείο ο δικός σας ρόλος είναι σημαντικός. Και βέβαια όχι μόνο ο δικός σας και των κρατών μελών και της βιομηχανίας. Χρειάζονται, χρειάζεται να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις κλειδιά με αποτελεσματικό τρόπο για να χτίσουμε την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω το ακριβές περιεχόμενο, τελικό περιεχόμενο του πρόγραμματος δράση για την άμυνα, αλλά μπορώ να σας δώσω μια ιδέα, μια γεύση, μια πρόγευση για την ακρίβεια αυτού. Να σας πω μερικά στοιχεία τα οποία είχαμε στο μυαλό μας. Ε, ε, πρώτο στοιχείο, πρώτος πυλώνας η καινοτομία και η έρευνα. Γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητά μας, θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Και σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Αν συγκρίνουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ, ειστερούμε. Χρειάζεται λοιπόν να ε, είμαστε πιο φιλόδοξοι. Όπως θα γνωρίζετε, έχουμε κάποιες ε, εντάξεις στον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς, ε, μερικές ε, δράσεις προετοιμασίας, προκατακτικές δράσεις, οι οποίες θα δίνουν ένα μήνυμα ότι η άμυνα είναι, βρίσκεται πλέον στον προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Είναι πολύ σημαντικό βήμα και είναι σημαντικό ε, επειδή πρέ, αυτές οι προκατακτικές δράσεις θα πρέπει να δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Γιατί θα πρέπει να αποδείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε για να φέρουμε καρπό. Και αν πετύχουμε σε αυτό, αν πετύχουν αυτές οι δράσεις και με σίγουρος θα πετύχουν, πρόθεση της Κομισιόν μάλλον είναι να ζητήσει στο επόμενο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο ένα ε, κονδύλι ειδικά για την ε, έρευνα σε θέματα άμυνας. Ε, αυτό θα το προτείνει η Κομισιόν. Τώρα βέβαια θα συζητηθεί με τα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο κλπ. Αλλά θα ήταν ένα μήνυμα για να δείξουμε ότι κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη. Από αυτή την πλευρά θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή που είναι σημαντικό για μας. Αυτός ο μελλοντικός ε, προϋπολογισμός αμυντικής έρευνας δεν θέλουμε, αν έτσι, δεν θέλουμε να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει αυτό που σημαίνει στα κράτη-μέλη. Θέλουμε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, αυτός ο προπολογισμό να προστεθεί στους προπολογισμού των κρατών μελών, όχι να μεταφερθούν κονδύλια από τους εθνικούς προπολογισμού ε, σε αυτό το πρόγραμμα. Δεύτερος ε, άξονας είναι ότι θα πρέπει να εστιαστούμε σε σημαντικά ε, ερευνητικά προγράμματα ε, τα οποία τα έχουμε ανάγκη, ε, για προϊόντα τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Δηλαδή θα συζητήσουμε με τη βιομηχανία, θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα δύο, τις ανάγκες με τις ικανότητες. Δηλαδή η έρευνα δεν είναι αυτός ο σκοπός, έρευνα για την έρευνα. Μετά, κίνητρα, οικονομικά κίνητρα. Τα ερευνητικά προγράμματα είναι ένα πράγμα. Χρειαζόμαστε όμως και οικονομικά κίνητρα στον τομέα της έρευνας. Για παράδειγμα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν. Είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα. Αλλά το βλέπουμε πολύ έντονα στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τις βοηθήσουμε να βρουν χρηματοδότηση στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος Γιούνκερ μίλησε για τη δημιουργία ενός ε, αμυντικού ταμείου, ταμείου άμυνας, για το μέλλον. Αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό από το ερευνητικό πρόγραμμα. Τώρα, συνεργαζόμαστε για να ε, ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα δράσης αλλά μία δυνατότητα, μία δυνατότητα λέω, είναι να δούμε το Ταμείο Γιούνκερ. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέματα άμυνας. Υπάρχει ένα ε, κανόνα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που λέει ότι ε, δεν είναι δυνατόν η άμυνα να αποτελέσει δικαιούχο δανείων. Οπότε εξετάζουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα και για τον αμυντικό τομέα. Δεν θέλω να προδικάσω την έκβαση. Δεν θα ληφθεί η ε, απόφαση αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αργότερα. Τελευταίος πυλώνας του πρόγραμματος δράσης είναι η εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά ε, ε, είναι πετυχημένη σε άλλους τομείς, γιατί όχι και στην άμυνα. Θα χρειαστούν τι να χρησιμοποιήσουμε τα ε, νομικά κείμενα που ήδη διαθέτουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κείμενο σε ό,τι αφορά τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας και το δεύτερο είναι η, η ονομαζόμενη οδηγία μεταφορών, μεταφοράς. Ε, δεν θέλουμε άλλα νομικά κείμενα. Εξετάζουμε τη χρήση αυτών των κειμένων, αυτής της νομοθεσίας. Ε, εξετάζουμε πώς έχουν εφαρμοστεί και ειλικρινά ε, θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί πολύ καλύτερα. Και προσπαθούμε, εξετάζουμε μάλλον, το πώς θα μπορούσαμε να ε, εφαρμόσουμε καλύτερα αυτά τα κείμενα, αυτή την νομοθεσία. Και η καλύτερη εφαρμογή μπορεί να γίνει είτε βέβαια με... Ε, <clears throat> με την γνωστή οδό της ε, ε, αστυνόμευσης ας πούμε αλλά μπορεί να γίνει και με κατευθυντήρες γραμμές γιατί <clears throat> ορισμένα από τα πράγματα που θεωρούσαμε ότι ήταν προφανή προφανώς δεν είναι ενδεχομένως θα μπορούσαμε λοιπόν να <clears throat> δημοσιεύσουμε κατευθυντήρες γραμμέ για την καλή εφαρμογή αυτών των νομοθετικών κειμένων. Αυτοί είναι οι τρει βασικοί πυλώνες του σχεδίου δράση για την άμυνα. <clears throat> Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση. Δεν έχει υιοθετηθεί, αλλά ακόμα και όταν υιοθετηθεί, δεν είναι το τέλος της διαδικασίας, αλλά η αρχή μιας διαδικασίας διαβούλευσης, στην οποία θα βέβαια θα συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για την ενημέρωση και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκρέχαμ για να μας μιλήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ. Νομίζω ότι είναι μια σαφής ένδειξη του πολύ στενού της πολύ στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας, ε, Εξωτερικών Δράσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Φεντερίκα Μουγερίνη επαναλαμβάνει ότι ε, έχει τους τρεις ρόλους ε, της, ε, είπα, προσώπου, της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επικεφαλής του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε εξ αρχής. Ο κύριος Μολενάρ είπε κάποια πράγματα για το επίπεδο φιλοδοξίας. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι οποιοδήποτε επίπεδο φιλοδοξίας και αν έχει κανείς θα χρειαστεί σίγουρα στρατιωτικές ε, δυνατότητες για να το επιτύχει γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρει. Και αυτό αυτό είναι ο ρόλο που έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα. Επίση, ε, ακούστηκαν κάποιε συγκεκριμένε προτάσει για δράσει. Ε, σε αυτό το τομέα ακριβώ θα επικεντρωθεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα και πολύ σύντομα να σας ε, περιγράψω, υπάρχουν πέντε σημαντικά πεδία. Καταρχάς, οι δυνατότητες άμυνας. Ε, είχα πει και, είπα και προηγουμένως ότι χρειάζεται κανείς ε, αμυντικές δυνατότητες για να επιτύχει το επίπεδο φιλοδοξίας του. Είναι κρίσιμη σημασία λοιπόν δεν έχουμε όλα τα είδη δυνατοτήτων που θα θέλαμε σε πληθώρα στην Ευρώπη δυστυχώ, Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να ενημερώσουμε, να αναθεωρήσουμε και να ενισχύσουμε ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μα για να καθορίσουμε δράσει προτεραιότητα, που είναι το σχέδιο ανάπτυξη δυνατοτήτων και ζητούμε την έγκριση βεβαίω των Υπουργών για να γίνει αυτό, ε, κάτι που θα, το, θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου στο Συμβούλιο. Ένα σημαντικός τομέας ε, ο οποίο, ωστόσο δεν είναι και πολύ ε, τραβηχτικός, πολύ ελκυστικός ε, για τα ε, ε, μέσα μαζική ενημέρωση είναι οι critical enablers. Οι δυνατότητε δηλαδή κατάρτιση, κατάρτισης, αξιολόγησης, δοκιμών. Είναι πολύ, σημαντικές αυτές, είναι πολύ σημαντικός αυτό το και υπάρχει τεράστιος κατακαιρματισμό και μάλιστα μεγάλη επικάλυψη στις προσπάθειες. Ο τρίτος ε, κλάδος πάνω στον οποίο θα δουλέψουμε είναι οι βασικές ε, στρατηγικές δραστηριότητες που θα είναι απαραίτητες για να ενισχύσουμε αυτό που λέγεται στρατηγική αυτονομία ή θα μπορούσε να ονομαστεί και ελευθερία δράσεων. Ε, να κάνω εδώ μια παύση και να υπογραμμίσω ότι εδώ δεν μιλούμε για, τη δημιουργία ενό οχυρού, μια Ευρώπη οχυρού. Προσπαθούμε η Ευρώπη να έχει τη δυνατότητα να δρά όταν χρειάζεται αυτόνομα. Είτε σε πολυμερείς, σε ε, ε, πολυμερή διεθνή μορφώματα ή και από μόνη της. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να το εξασφαλίσουμε αυτό και δουλεύουμε από κοινού με την Γενική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση GROW και τη βιομηχανία. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την, ε, τις τεχνολογικές εξελίξεις, ε, τις βιομηχανικές ε, εξελίξεις, τα προσόντα. Περνάμε τώρα στον τέταρτο τομέα. Η τεχνολογία και η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντικός τομέας. Αν δεν επενδύσουμε στην έρευνα και την τεχνολογία σήμερα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις δυνατότητες του αύριο. Και όταν λέω αύριο εννοώ σε 10-15 χρόνια. Επίσης κάτι άλλο σημαντικό και συμφωνώ με τον κύριο Ντελσό απολύτως, ό,τι και αν γίνει σε επίπεδο ε, ερευνητικών προγραμμάτων για την άμυνα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρόσχημα για τα κράτη-μέλη για να σταματήσουν να πιέζουν και να επιταχύνουν ε, τις εθνικές επενδύσεις στην έρευνα για την άμυνα. Αυτό είναι κρίσιμη σημασίας και συμφωνώ μαζί του, δεν υπάρχει, δεν αντικαθιστούμε εδώ κάτι, ούτε υποκαθιστούμε. Είναι ενίσχυση της γενικότερης δυνατότητας επένδυσης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι 7 φορές λιγότερη συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και τέλος, πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ώστε να γίνει πιο ελκυστική η συνεργασία. Η παγκόσμια συνεργασία λέει ότι θα πρέπει να γίνει ο κανόνα η συνεργασία. Ε, αυτό μάλλον ε, πιο εύκολα το λέει κανεί παρά το κάνει. Όπω είπε όμω και ο Πιέρ Ντελσό, προσπαθούμε να ε, βρούμε κάποια κίνητρα. Μπορεί να είναι δημοσιονομικά, μπορεί να είναι εξαιρέσει από τον ΦΠΑ, ελαφρύνσει φορολογικέ για προγράμματα τα οποία μπορεί να είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα. Μπορεί να υπάρχουν και χρηματικέ διευκολύνσεις. Εδώ βεβαίω δεν θέλω να μπερδευτούμε με αυτό που περιέγραψε ο Πιάκ Ντελσό. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ένα είδος μηχανισμού που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη κάποια από τα δικά τους κονδύλια, μπορεί να είναι και ένα μείγμα ε, δημοσίων και ιδιωτικών ε, επενδύσεων, γιατί βεβαίω πάντα υπάρχει το πρόβλημα του προπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί κάποια κρατημέλη να έχουν ας πούμε, την ίδια απέτηση, το ίδιο, την ίδια ανάγκη στα, στην ίδια, την ίδια χρονική στιγμή και να μην υπάρχει ο, ο προπολογισμό για να γίνει αυτό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υπάρξει ένα μηχανισμό για να ε, προσπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Και επίση, ε, τμήμα αυτή τη δουλειά είναι και το να δούμε όχι αυτό που ονομάζουμε ε, εξάμεινο άμυνας. Ε, έχουν γίνει διάφορες αναφορές βεβαίως και είναι αρκετά χρήσιμο. Αλλά αυτό, αυτή η συντονισμένη αιτήσια αναθεώρηση που θέλουμε να υπάρχει ένας τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα προσπαθήσουμε τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμίσουν τα σχέδια άμυνας που έχουν έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη πίεση ομοτήμων που δεν είναι ιδιαίτερος παρούσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να μετακινηθούν λίγο από τους συλλογικούς εθελούσιους στόχους που είναι ανούσιοι ουσιαστικά σε κάτι πιο μεμονωμένο, επιμέρους και ίσως πιο πολιτικά δεσμευτικό. Αυτό, αυτές είναι κάποιες από τις ε, ιδέες για τις οποίες θα κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις για δράση. ώστε να συμπεριληφθούν ε, σε αυτό το σχέδιο το εφαρμοστικό για την ε, άμυνα και την ασφάλεια. Και σε αυτό μπορώ να ολοκληρώσω την, με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ. Τρεις συντονιστές έχουμε εδώ από τις πολιτικές ομάδες, οπότε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά, βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ τους κυρίους για τις παρεμβάσεις τους. Μου άρεσαν αυτά που άκουσα. Εμείς ως ΕΛΚ συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας και τις προσπάθειες που κάνετε για να ενισχύσετε την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι από την πλευρά του Κοινοβουλίου δεν ε, λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα ψηφίσματα, ας πούμε, όπως του 2013, του 2015. Δεν εφαρμόζονται, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και βεβαίως ε, υπάρχει ε, έλλειψη στην ε, εφαρμογή. Από, την, ε, από το τέλος του Αυγούστου είπα ότι εκπρόσωπος μιλά για την θέση της Ευρώπης και μιλά για την εφαρμογή. Βεβαίως αυτό δεν συνάδει με τις δικές μας ε, απαιτήσει που έχουμε ήδη παρουσιάσει και τις οποίες έχουμε συμφωνήσει και στην Λευκή Βίβλο για την άμυνα και την ασφάλεια, κάτι που το ζητούμε εδώ και καιρό. Και επίση, δεν παίρνει τόσο σοβαρά υπόψη της την ε, παγκόσμια στρατηγική, στην οποία αναφέρεται στη σελίδα 45, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, ε, μια τομεακή στρατηγική για τον ορισμό του επίπεδου φιλοδοξίας, τα καθήκοντα, οι απαιτήσει και οι δυνατότητες, καθώς επίσης και οι προτεραιότητες. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε παρά την πολύ σαφή αναφορά που γίνεται εδώ για τη δημιουργία μιας ε, τομεακής αμυντικής στρατηγικής γιατί ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο εφαρμογής. Ε, η Κομισιόν επίσης πάνω σε τι ε, δουλεύει, τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα, το οποίο τέλος Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμο. Σας ρωτώ, ρωτώ βεβαίως και τα κρατημέλη, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας στο σχετικά με το PSK και τη, που είχε προταθεί από το 2014. Ήδη από τις αρχές του 2014 υπήρξε παρουσίαση του σχέδιου αυτού και βεβαίως έτυχε μεγάλης υποστήριξης. Τελικά τι έγινε με το σχέδιο αυτό, που βρίσκεται. Δεν νομίζουμε ότι έχουν γίνει πολλά. Οπότε τώρα μιλούμε για, την, ε, ε, για, μια, για ένα νέο σχέδιο, την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου, χωρίς να έχουμε εφαρμόσει το παλαιό. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιες σκέψεις για το πώς προχωρούμε. Ε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταλήξουν τελικά να εφαρμόσουν αυτά που συμφωνούν. Υπάρχει και η ανακοινωθήσα ήδη πράσινη βίβλος για τους οδηγικούς ε, πόρους και, το, και, το, και ο δικός χάρτης επίσης για την ε, ασφάλεια και για τη δημόσια τάξη. Τι γίνεται με αυτό. Επίσης τα θέματα χρηματοδότησης. Ε, κάναμε πολλές ε, συζητήσεις και σήμερα το πρωί για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, για την έρευνα, για την άμυνα που προωθείται με ένα πιλωτικό πρόγραμμα ήδη από το 2015 και για το 2016. Στο περιθώριο αυτό το Κοινοβούλιο στην εφαρμογή της απόφασης ε, του 2013 είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή. Μιλήσατε λίγο για το 2017, για την ε, ε, έγκριση της Επιτροπής Περιπολογισμού, για τα απαραίτητα κονδύλια, για την έρευνα για την άμυνα, που βεβαίως ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση, η οποία όμως είχε ευτυχές τέλος. Δυστυχώς, δεν καλύψατε όμως τη δική μας, ε, το δικό μας αίτημα για την ανακοίνωση της Κομισιόν του, ε, που θα δημοσιευθεί τώρα το, που δημοσιεύθηκε συγγνώμη φέτος το καλοκαίρι. Βεβαίω είπαμε ότι εδώ δεν υπάρχει υποκατάσταση των εθνικών ε, προσπαθειών. Μιλάμε για ενίσχυση αυτών, για μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. για να βελτιώσουμε δηλαδή το τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Ίσως όμως ε, αν είχαν γίνει όλα αυτά πιο πριν να μην είχε χρειαστεί να κάνουμε την ε, συζήτηση αυτή. Αν κάνουμε την ίδια συζήτηση όμως το 2017 και το 2018 Καλό θα ήταν να δούμε και, τις, ε, και την έγκριση που μπορούμε να πάρουμε από την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού. Με την, ε, υπήρξε και συμβασμός βεβαίως, γιατί ζητούμε παρκείς, βιώσιμες πηγές χρηματοδότησης και λυπούμεθα που τα τρία, το, ποσό των, το ποσό για τα τρία χρόνια δυστυχώς μειώθηκε. Τα κράτη-μέλη δεν ξέρω κατά πόσο θα δώσουν νέα ε, κονδύλια για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν μια αναθεώρηση και να απαντήσουν στο ερώτημα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, ε, Άμυνας πώς μπορεί να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με κατάλληλο τρόπο για την επόμενη προγραμματική περίοδο και το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα κάποια ερωτήματα εκκρεμή. Τρία χρόνια μετά την Σύνοδο Κορυφή για την Άμυνα, μπορώ να διαπιστώσω ότι τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν έχουν... Ε, δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη τα μέτρα για την, ε, ε, για την άμυνα και την ασφάλεια. Υπάρχουν κάποιοι που επωφελούνται από αυτό. Ο Αλμπαγκδάτη, ας πούμε, του α, Ισλαμικού κράτους ή κάποιοι άλλοι, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το επιτρέψουμε αυτό να συμβαίνει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόνιντ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, είμαι ο μόνος από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, που θα έπρεπε να παρουσιάζει αυτή τη θέση. Ε, αλλά είμαι από την Αυστρία και πρέπει να το αναφέρω αυτό σήμερα, όπως έχω κάνει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Η Αυστρία είναι ουδέτερη χώρα ουδέποτε ναι, είμαστε ανέκαθεν είμαστε ουδέτεροι και μη ρωτάτε απέναντι σε ποιον. Εμείς έχουμε κάνει λοιπόν μερικά πρώτα δηλάβηματάκια ματάκια προς το ΝΑΤΟ και σε σχέση με τη βασική μας αντίρρηση κατά της οποιασδήποτε μορφής στρατιωτικοποίησης. Η κατάσταση βέβαια μεταβάλλεται στην άμεση γειτονιά μας, οπότε μάλλον πρέπει να ξαναδούμε και τη δική μας θέση και να ξανασκεφτούμε το δόγμα ουδετερότητας της Αυστρίας. Πέραν αυτού πρέπει να προσθέσω ότι με το Brexit πρώτων πυλών και την ε, Μεγάλη Βρετανία να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άμεσο μέλλον. Υπόθηκε και το πρωί. Η Βρετανία είναι πυρηνική χώρα. Και έχει πολύ δυνατό στρατό. Είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ήταν σημαντικό αυτό για όλες τις όψεις της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Θα χάσουμε λοιπόν, αν και ελπίζουμε να μην χάσουμε τελείως τη συνεργασία τους. Θέλω επίση να πω το εξή Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων θα μπορούσε και αυτό να είναι μια πηγή εισοδημάτων για την ε, βιομηχανία της άμυνας αλλά λέτε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχω και εγώ κάποιε αμφιβολίε για το αν αυτή θα ήταν καλή λύση για τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το ΕΦΣΙ δημιουργήθηκε προκειμένου να τονώσει, να δώσει μια όθηση στις, ε, στα δύναμα ποσοστά ανάπτυξη της Ευρώπης. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος πως η έρευνα σε θέματα άμυνας θα συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο κατεπηγόντως χρειαζόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Επίσης αναφέρατε ότι κοιτάζετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς και πώς εφαρμόζονται τα σχετικά με την άμυνα. Δεν είμαι βέβαιος τι εννοούσατε. Εάν θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λέζινγκ της Γκουέ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ πολύ τις ε, παρουσιάσεις ε, που έγιναν και συμφωνώ με, τους, με τα σχόλια του συναδέλφου. Για αυτά που είπε ο συνάδελφος Φρόιντ να πω ότι δεν είμαι μόνο απογοητευμένη, ότι είναι τόσο λίγοι οι σοσιαλιστές σήμερα εδώ, αλλά γενικώ ότι είναι τόσο πολλοί οι ευρωβουλευτές σήμερα εδώ στην υποεπιτροπή μας για να... και συζητούμε μεταξύ μας ουσιαστικά τα πολύ σημαντικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέματα που έχουν ε, να κάνουν και με την ασφάλεια των πολιτών αλλά και με την κατεύθυνση που θέλει να πάρει η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω ότι συμφωνεί και ο συνάδελφος Γκάλερ Σπάνια υπάρχουν τέτοιε συμμαχίε εδώ στην Επιτροπή. Μάλλον ε, θα αλλάξει πολύ σύντομα αυτό, το φαντάζεστε. Οπότε θέλω να θέσω το ερώτημα, το είπε και ο κύριος ε, Φρόιντ. Η χρήση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για την έρευνα για την άμυνα. Εκεί θα ήθελα λίγο πιο λεπτομερείς απαντήσεις. Η παράγραφος ε, 41.1 λέει σαφώς ότι τα μέσα για τα προγράμματα ασφάλειας και άμυνας ε, δεν θα προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Οπότε θέλω να θέσω το ερώτημα, υπάρχει κάποια νομοθε... Ε, δεσμευτική νομοθετική γνωμοδότηση ή το Κοινοβούλιο απλώς μπορεί με ψηφοφορίες να τα αλλάζει αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δημοκρατικό αυτό, οπότε αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε πότε σκέφτεστε να ενημερώσετε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ερμηνεύετε τις ε, διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας με αυτόν τον τρόπο. Ίσως αυτό να επηρεάσει και τις, ε, ε, τις αποφάσεις που θα πάρουν για τις επόμενες ευρωεκλογέ. Επίσης, ε, μιλήσαμε γενικά για διάφορα θέματα, για τη βελτίωση των δυνατοτήτων κλπ. Αρκετά ενδιαφέρον είναι να μιλήσουμε ίσως και για πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Ας πούμε, ο φιλόδοξος αυτός στόχος για, τις, για τη βελτίωση των δυνατοτήτων που, μιλήσατε, που είπατε και εσείς, ο ορισμός επίσης το, για, το διάφορο, για το φάσμα των δυνατοτήτων που έχουμε από αέρος, τις χερσαίες δυνάμεις, τις αεροπορικές δυνάμεις κτλ. και πώς αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες. Είπαμε ότι είναι φιλόδοξος ο στόχος αυτός, από τον οποίο απέχουμε βεβαίως πόρο ακόμη ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ξέρω, θα, θα ήθελα να μου πείτε κάποια αριθμητικά στοιχεία για τις επιπλέον ίσως ε, επενδύσεις που θα ήταν απαραίτητες. Και άλλο ένα ερώτημα για το ε, θέμα των αιτιών ε, των, της αντιμετώπισης των αιτιών της, των διώξεων και της δυνατότητας αντιμετώπισης αυτής. Ποιοι είναι δηλαδή οι λόγοι ακριβώς, γιατί πρέπει, όχι γιατί αναγκάζονται να φύγουν, γιατί πρέπει να φύγουν. Ένα μεγάλο κομμάτι της ε, πολιτικής ε, γειτονίας ε, και πολλές χώρες στην περιοχή βυθίζονται στον, στον όλεθρο και στις συγκρούσεις. Και υπάρχουν και διάφορες συνθήκες, συμφωνίες σύνδεσης με τις γειτονικές χώρες για την ε, δημιουργία ελεύθερων ε, ζωνών ε, εμπορίου. Εγώ πάντα με μεγάλη έκπληξη βλέπω ότι και ο κύριος Μπροκ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, λέει πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξανασκεφτεί την πολιτική εμπορίου της. Αλλά σπάνια ακούω περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν διάφορες ε, μελέτες που λένε ότι αυτές οι, ε, αυτή η πολιτική προκαλεί πολλά προβλήματα. Ε, τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη και αν ναι, ποιες είναι οι προσπάθειες που γίνονται για να, λύσουν, να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Επίσης, η Λευκή Βίβλος έχει καταγραφεί ως αίτημα και εγώ ήθελα να το τονίσω αυτό και να θέσω και σε εσά το ερώτημα. Η ευρωπαϊκή ε, στρατηγική πώς πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη. Θα υπάρξει μια λευκή βίβλος και θα είναι επίκαιρη. Θα περιλαμβάνει τις ε, διατάξεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας για την ατζέντα που έχουμε προωθήσει και η οποία θα πρέπει να μπει σε ε, διαδικασία έγκρισης το 2016. Ευχαριστώ. Very indeed. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση. Τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Grow. Ε, τι είδου ανάλυση slot πρέπει να κάνουμε για να εντοπίσουμε τους μηχανισμούς και τους ε, τομείς στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε. για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι προσπάθειές μας θα έχουν προστιθέμενη αξία. δεδομένου ότι η κατάσταση ε, της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δυσχερής. Με την ίδια σειρά, έτσι. Καταρχήν ο κ. Μολενάρ, μετά ο Γενικός Διευθυντής, ο, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κ. Δελσό και μετά ο κ. Μέρ. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Τα καταγράφουμε κύρια ερώτηση που προκύπτει από ό,τι βλέπω είναι για τη λαϊκή Βιβλό. Μεταξύ των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου αναφερόταν και ελήφθη υπόψη όταν μιλούσαμε για τη σφαιρική στρατηγική, τη διεθνή αυτή στρατηγική της Ένωσης. Προσωπικό σχόλιο τώρα, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω πρώτο είναι να μην κρίνουμε το βιβλίο από το εξώφυλλό του. Λευκό βιβλίο μεν, αλλά το θέμα είναι τι περιεχόμενο θα έχει, τι θέλουμε δηλαδή να είναι το ζουμί. Ίσως να μην είναι αρκετά έντονη η δήλωση και πραγματικά αυτό που θέλουμε είναι τα αποτελέσματα να είναι απτά, να επικεντρώνονται στην χειροπιαστή δράση. Ταυτόχρονα, αν σκεφτείτε σε τι ύψο φιλοδοξιών έχουμε φτάσει, κάτι που θα ανοίξει νέα πεδία εργασία για μα ή τέλο πάντων θα υποστηρίξει κάποιε γραμμέ εργασία που ήδη έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν, θα δοθεί μια πιο συστηματική και ε, μεθοδική διάσταση στις δραστηριότητες της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, εκεί πρέπει να γίνουμε πιο αντιδραστικοί και πιο, να αντιδρούμε μάλλον πιο γρήγορα και να κινούμαστε πιο γρήγορα και σε ό,τι αφορά τις μάχημες ομάδες, μονάδες και την οικοδόμηση δυνατοτήτων στα εργαλεία ασφάλειας και ανάπτυξης ταυτόχρονα αλλά και προστασίας εξωτερικός και εσωτερικός. Πρέπει δηλαδή η ασφάλεια και η άμυνα στην Ευρώπη να πάρουν τέτοιε διαστάσει που να επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τι πραγματικέ απειλέ που αυτή τη στιγμή βαρύνουν την Ευρώπη. Προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα βασιζόμενοι στι προτάσει τη σφαιρική στρατηγική. Τι προτάσει σα, λοιπόν, για να είμαστε όσο δυνατόν πιο φιλόδοξοι, τι ε, καταγράφουμε προσοχή. Αλλά πραγματικά μην κρίνετε το περιεχόμενο του βιβλίου από το εξώφυλλό του. Υπάρχουν κάποιοι στρατηγικοί προσανατολισμοί που ελπίζουμε να επικρατήσουν ε, για τα ερχόμενα χρόνια. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και κοιτάζουμε να διερευνήσουμε αυτό το πεδίο. Ε, αυτή είναι ακριβώ τη φάση που βρισκόμαστε. Αυτή νομίζω ήταν μια από τι βασικέ παρατηρήσει. Τώρα για τον Brexit και τον αντίκτυπό του. Δύσκολο εγώ να σχολιάσω για το τι ακριβώ αντίκτυπο θα έχει. Φυσικά είναι ένα παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη στι συζητήσει. Είναι και ένα θέμα που συζητιέται ευρέω και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε εμεί αυτή τη χρονική στιγμή πέραν από όσα λέγονται σε επίπεδο κοινή γνώμη, αλλά σίγουρα μα απασχολεί στα πλαίσια αυτή τη ενεξελίξη συζήτηση. Δεν. Δεν ξέρω ποιον τίτλο θα δώσουμε, ώστε να μην είναι αρκετά υπεροπτικός. Ε, προσπαθούμε να διαλέξουμε κάτι μετροπαθές, σχέδιο ή πρόγραμμα υλοποίηση εφαρμογή, κάτι με περισσότερη εγκροέτεια. Ευχαριστούμε, Διευθυντά Ντελσό, για το πρόγραμμα υλοποίησης. Τα έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές αυτό το σώμα και εσείς όντως είχατε πολλή βούληση και πολύ ε, δράση για να είμαστε φιλόδοξοι εδώ. Όμως εκτός του Κοινοβουλίου δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βλέπετε ότι κάποια κράτη-μέλη μάλιστα έχουν ε, διαφορετική διάθεση, έχουν αποστείλει και σχετικές επιστολές. Ε, Πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο μάλιστα έχουν. Η άμυνα είναι κάτι, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται διαφορετικά πλέον από τι κυβερνήσει και έχει διαφορετική θέση στι προτεραιότητε των κυβερνήσεων στι διαπραγματεύσει. Και εγώ πραγματικά απογοητεύτηκα και αισθάνθηκα μεγάλη ε, ματέωση, αλλά βλέπω να υπάρχει αλλαγή στη στάση των κρατών μελών. Και είναι κάτι που το ενθαρρύνουμε και ελπίζουμε θα οδηγήσει κάπου. Δεύτερη γενική παρατήρηση. Ο τομέα τη άμυνα είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Εάν δείτε του αριθμού, και επανέρχομαι στην ερώτησή σα, Πρόεδρε, έχουμε αριθμού για το ποιοι απασχολούνται στον τομέα τη άμυνα, ε, ποιο είναι ο κύκλο εργασιών. Είναι ένα σημαντικό τομέα, κλάδο για την Ευρώπη. Όμω, ε, εκεί δεν δραστηριοποιούνται μόνο μεγάλε επιχειρήσει, αλλά και πολλέ μικρομεσαίε όλων των κρατών μελών. Και ίσω να μην σα αρέσει η άμυνα αυτή καθεαυτή, όμω είναι πολύ ο κόσμο που δουλεύει σε αυτόν τον κλάδο και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να του βοηθήσουμε είναι και αυτή μια από τις πτυχές ε, που θέλαμε να, μας, να μελετήσουμε καλύτερα. Δεύτερο στοιχείο, και συμφωνώ μαζί σας κύριε Γκέλλερ, πρέπει, μάλλον δεν θέλουμε ο νέος οργανισμός άμυνας, και θα μιλήσω για αυτό, δεν θέλω να γίνει σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο φορτωμένο με 35 χριστουγεννιάτικες μπάλες μέτρα που να μην οδηγήσουν πουθενά. Θέλουμε ένα περιορισμένο αριθμό δράσεων για να πετύχουμε και χειροπιαστά αποτελέσματα. Ιδάλω, άλλο ένα έγγραφο που θα περάσει τα γραφεία τη Επιτροπή θα εγκριθεί και δεν θα κάνει τίποτα, θα είναι και αυτό. Θέλουμε κάποιε βασικέ δράσει που αυτέ να υλοποιηθούν. Υπό αυτή την έννοια, το πρόγραμμα έρευνα είναι κάτι που είναι άκρο σημαντικό για μα. Κυρία Λέζιν, για να επανέλθω στην ερώτησή σα για τη νομική βάση. Σε κάποιο βαθμό η συζήτηση αυτή έχει ήδη γίνει στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων. Βεβαίω, ο προπολογισμό ε, του 2017 δεν έχει ακόμα εγκριθεί επισήμω, αλλά φάνηκε και από τι συζητήσει και από τη σκοπιά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σαφέ ότι. Σα λέω ποια είναι η θέση μα, δεν σα λέω τι θα γίνει, δεν προδικάζω. Ότι τέτοιο ερευνητικό πρόγραμμα ε, προβλέπεται το κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει βεβαίω αν είναι σωστό ή όχι κάτι τέτοιο να γίνει. Αλλά από τη δική μα την πλευρά είναι εφικτό. Και άλλε δύο σύντομε παρατηρήσει για το ΕΦΣΥ. Και πάλι δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει. Δεν ξέρουμε αν θα πετύχει. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα να επικεντρωθούμε μόνο στην έρευνα αυτή καθεαυτή. Είναι τι θα κάνουμε με την έρευνα. Έρευνα μπορεί να γίνεται. Αλλά πρέπει κάτι να μπορούμε να φτιάξουμε από αυτήν. Δηλαδή προϊόντα ε, που να έχουν προκύψει από τι ερευνητικέ προσπάθειε. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε τι ανάγκε μα. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθεί και χρηματοδότηση. Οι μικρομεσαίε δεν βρίσκουν εύκολα χρηματοδότηση. Ιδίω στον τομέα και τον κλάδο τη άμυνα. Ε, ισχύει περισσότερο σε άλλους ίσως τομείς, αλλά στο δικό μας το κλάδο είναι πραγματικά πολύ ε, σημαντικό στοιχείο. Κοιτάζουμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε κάποια διέξοδο, κάποια πρόσβαση σε αυτό το, ε, σε αυτό επίπεδο και στις μικρομεσαίες για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν, για τις δημόσιες προμήθειες. Εδώ υπάρχει σχετική οδηγία. Ε, εγκρίθηκε πριν από λίγα χρόνια από το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Ε, αυτή η οδηγία ζητά κυρίω από τα κράτη-μέλη να είναι περισσότερο ανοιχτά στι δημοσιε προμήθειε του τομέα της, του κλάδου της άμυνας. Δηλαδή, όχι να τα κάνουν όλα δημόσια, ε, δημοσίω, αλλά για τον στρατιωτικό εξοπλισμό κάποια πράγματα να είναι ανοιχτά. Δηλαδή, το κείμενο υπάρχει στην νομοθεσία του συνήθω, αλλά δεν το εφαρμόζουν αναγκαστικά. Οι υποχρεώσει του ε, είναι πολύ λίγε και είναι περιορισμένε πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σε επίπεδο οδηγία, γιατί θα ήταν πολύ περίπλοκο, αλλά θέλουμε να κοιτάξουμε προσεκτικά την οδηγία και προτού εφαρμοστεί επιτόπου από τα κάτι μελη θέλουμε να ξέρουμε ότι θα τονώσει τον ανταγωνισμό και ότι θα είναι πιο ανοιχτή αγορά. Διότι θα είναι σημαντικό για όλε τι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην αγορά, για τι μεγάλε και τι μικρομεσαίε, να υπάρχει διασυνοριακή ε, πρόσβαση. Ξέρουμε ότι η άμυνα είναι ένα θέμα ευαίσθητο, αλλά γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να σα μιλήσουμε και να σα διαφωτίσουμε για αυτό το θέμα. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι είναι μια σημαντική βιομηχανία, ένα σημαντικό βιομηχανικό κλάδο τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, πράγματι. Τρίτο, ο κύριο Μιουρ. Επιτρέψτε μου μόνο μια παρατήρηση. Καλωσορίζουμε την ομάδα επισκεπτών παρατηρητών μάλλον. Παρακαλώ όμω καθίστε και θα σας παρακαλέσω όποτε θελήσετε να βγείτε από την αίθουσα κάντε το όταν θα ολοκληρώσει ο επόμενος ομιλητής μας. Είναι πολύ ενοχλητικός ο θόρυβος και σας καλωσορίζουμε με θερμά αλλά ελπίζουμε να έχετε άριστη διαγωγή. Διότι όσο περισσότεροι πηγαίνουν έρχονται, τόσο πιο δύσκολο να μιλήσει κανεί. Εάν θελήσατε λοιπόν να εξέλθετε ε, μετά, παρακαλώ να το κάνετε μετά τις παρεμβάσει. Um, uh, fairly... Θα είμαι σύντομο. Μιλώντας σε προσωπικό επίπεδο, αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση που αυτή η στρατηγική δεν είναι μια λευκή βίβλος. Αυτό όμως που είναι σημαντικό όπως είπε ο κ. Μολυνάρη είναι το περιεχόμενο και όχι ο τίτλος. Γιατί τελικά η Κομισιόν, η, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ό,τι και να κάνουν δεν θα αλλάξουν την κατάσταση η άμυνα είναι αρμοδιότητα εθνική και η εφαρμογή του προγράμματος θα είναι τελικά εθνική ε, αρμοδιότητα και επιλογή. Είχαμε δύο-τρεις ερωτήσεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, για την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος. Να σας πω. το πειρατικό πρόγραμμα θα μας οδηγήσει σε ε, ε, προκαταρκτικές δράσεις. Είναι κάτι καινούριο. Ε, είναι χαρτογράφητα νερά. Ο λόγος που υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα είναι να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας. Είναι κάτι μικρό. Δεν είναι τρομακτικά απαιτητικό, οπότε είναι μια, ένα καλό σημείο κίνησης τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Και οι προκατατικές δράσεις θα είναι το επόμενο βήμα έτσι ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, έρευνας για την άμυνα στο επόμενο μεσοπρόθεσμο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν θα είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή, αλλά πάντως Πρέπει να δούμε πώς θα οργανωθούμε για να δώσουμε αποτελέσματα και με τους πόρους και με το κατάλληλο προσωπικό που χρειαζόμαστε, την τεχνογνωσία. Έτσι θα διαρευνήσουμε το τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Ε, και ασφαλώς θα ρωτήσουμε και τα κράτη-μέλη τι περιμένουν από, την, από τον οργανισμό μας ε, τα επόμενα χρόνια. Αναφερθήκατε στην ε, ασφάλεια προμηθειών, προμήθειας, στην ασφάλεια ανεφοδιασμού. Για να λειτουργήσει αυτή η ασφάλεια ανεφοδιασμού χρειάζεται δέσμευση. Και ακούμε τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αρκετή δέσμευση. Γιατί ε, αν έρθει ο κόμπος το χτένι θα χρειάζεται να έχουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται όταν το χρειάζονται ακριβώς, όχι αργότερα. Οπότε αυτή τη στιγμή η ασφάλεια ανεφοδιασμού μας ξεπερνάει. Τώρα κύριε κυρία Λέσσινγκ ρώτησε πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δεν γνωρίζουμε και κανείς δεν γνωρίζει νομίζω. Αλλά να το γυρίσω ανάποδα. Δεν είναι ότι τα κράτη-μέλη όλα μαζί δεν επενδύουν αρκετά στην άμυνα. Είναι 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, είναι τα μισά από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά δεν είναι και μικρή επένδυση. Το πρόβλημα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα υστερεί πάρα πολύ. Επενδύουμε το 50% των όσων επενδύουν οι Πολιτείες αλλά το αποτέλεσμά μας είναι 15% του αποτελέσματος που ανελαμβάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το 60% των επενδύσεων πηγαίνει σε προσωπικό. και δαπανούμε το 20% των όσων δαπανούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για εξοπλισμό. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι ότι μόνο ότι επενδύουμε λίγα, είναι ότι δεν παίρνουμε και επαρκή αποτελέσματα, δεν αποδίδουν επαρκώς οι επενδύσεις μας. Οπότε θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επενδύουν με πιο έξυπνο τρόπο. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάλλο, θέλετε το λόγο, είναι ικανοποιητική η απάντηση. I'm fine. I'm... Ε, δεν πήρα απάντηση. Τι θα γίνει με το πρόγραμμα ε, του Ιανουαρίου 2014. Σε ποιον την είχατε απευθύνει αυτήν την ερώτηση. Sorry, sorry. <laughs> No, I mean it was... Ο κ. Ποπόφσκι το είχε παρουσιάσει. Τώρα δεν ξέρω ποιο από τους παρόντες είναι πιο κοντά σε αυτό το θέμα. Ε, ο κ. Ποπόφσκι ήταν, ε, ανήκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής οπότε ε, ο λόγος στον κ. Μολυνάρ. Προσπαθώ να το θυμηθώ. Το πρόγραμμα εφαρμογή του 2014 Ε, το έχουμε αναφέρει στα συμπεράσματα και, τα, και παρακολουθούμε. Ε, κύριε μη, μη διακόπτετε. Σας δώσω το λόγο. Ε, ε, έχουμε τα συμπέρασματα του 2013 και του 2015, είναι σημαντικά, παραμένουν σε ισχύ. Αν τώρα χρειάζεται να παρακολουθήσουμε κάτι σε αυτά τα συμπεράσματα θα το παρακολουθήσουμε. Ε, τώρα ε, περνάμε στο επόμενο στάδιο βέβαια, αλλά πράγματι δεν πρέπει να ξεχνάμε και το προηγούμενο. Θέλετε ξανά το λόγο. Ωραία, σε ευχαριστώ. Κλείνουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ εκ μέρου σα και τους ε, τρει ε, ομιλητέ. Ε, είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε. του επόμενου μήνε, τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ παραμείνετε όμως, γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα στην μέση διάταξη. Ladies Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Υπάρχει ένα ακόμη σημαντικό και πολύ ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διαταξής μας, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σοβαρό από τα προηγούμενα, ένα θέμα που θα το χαρακτήριζα κάπως ε, συντομευμένο. Θέλαμε να έχουμε κάποιες τεχνικές συστάσεις για την επερχόμενη επισκεψή μας στην Ουκρανία και ο αρχικός σκοπός ήταν να επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και ορισμένα σημεία στην Ανατολική χώρα. Όμως, θα είναι κάπω προβληματική η διεξαγωγή μια τέτοια επίσκεψη λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται και τη κατάσταση ασφάλεια εκεί. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτήν την ενημερωτική σύνοδο για την ασφάλεια και την κατάστασή της στο Κίεβο προφανώ, αλλά ε, μπορεί να έχουμε εκπλήξει ε, μέχρι τότε και σίγουρα στην Ανατολική Ουκρανία ε, ο σκοπός της αποστολής είναι να ξεκινήσει 1η Νοεμβρίου το βράδυ και ο κύριος Αντριάνο Μάρτιν είναι προσκεκλημένος μας, Αντριάνο Μάρτινς ο οποίος είναι τμήματάρχης, υπεύθυνο για την ε, διμερή διάσταση της Ανατολικής Γειτονίας στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε αυτή λοιπόν τη φάση και εν ώψη της επίσκεψης της αντιπροσωπείας ΕΝΤΕ στην Ουκρανία θα θέλαμε να συζητήσουμε την κατάσταση της ασφάλειας την Ουκρανία εκ των προτέρων. Κύριε Μάρτινς, έχετε το λόγο. Όπως γνωρίζετε, η ασφάλεια δεν έχει επανεγκατασταθεί στην Ανατολική Ουκρανία. Ε, ο Οργανισμός των Εθνών ε, έχει καταγράψει 9.640 νεκρούς και 22.400 τραυματίες από την αρχή της κρίσης. Ε, και τα θύματα αυξάνονται κάθε μέρα περνάει. Αυτή η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία μας αναγκάζει να κάνουμε άλλη μια έκκληση ε, στις όλες τις πλευρές να βρουν μια μόνιμη λύση που θα ε, σέβεται την ενότητα, την ε, εδαφική ακαιρεότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Η συμφωνία του Μίνσκ είναι το βασικό εργαλείο για την επίλυση των διαφορών. Η ασφάλεια και οι πολιτικές προσπάθειες συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες εστιάζονται στην υιοθέτηση ενός οδικού χάρτη ε, ο Γερμανός και ο Γάλλος προς εξωτερικών το Σεπτέμβριο βρέθηκαν στο Κίεβο και αναφέρθηκαν σε μια σειρά τριών βημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολλά πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η συμφωνία του Μίνσκ να εφαρμοστεί καθ' ολοκλήρια. Σε ό,τι αφορά την ανακοχή ε, Πρόσφατα ε, είδαμε μία ακόμα προσπάθεια να ηρεμήσει η κατάσταση κατά μήκο τη γραμμή επαφή. Ε, οι παραβιάσει τη ανακοχή ε, έχουν μειωθεί, αλλά παρόλα αυτά είναι καθημερινές σε ό,τι αφορά το σχέδιο αποσύνδεσης. Ε, η ομάδα εργασία για θέματα ασφάλειας μετά από τρεις ε, μήνες, ε, στις 21 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε και υπογράφηκε και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία και από εκπροσώπους των διαφόρων περιοχών της επαρχίας του Ντονέτσκ και προβλέπει αυτό το σχέδιο την δημιουργία ε, ζωνών και την απομάκρυνση των δυνάμεων, ε, στρατικών δυνάμεων τη μια και από την άλλη μεριά. Ξεκινάμε με τρεις πολιτικές ζώνες, Στανίτσια, Λοράτσκα και Ζολότμπουφ, Καθώ επίσης και το Πετρίσκι στη, στον, στην περιοχή του Ντονέτσκ. Ε, έχει επιτευχθεί πρόοδο στις δύο πρώτες, ε, αλλά ο, ο ΑΣΕ, η ομάδα που κάνει το monitoring, δεν το έχει επιβεβαιώσει. Ε, διότι η δραστηριότητα της ομάδας παρακολούθησης ε, βρίσκει εμπόδια και από τις δύο πλευρές. Ε, αντιμετωπίζουμε σημαντικές, σημαντικά προβλήματα στην δουλειά μας. Μάλλον ο ΑΣΕ αντιμετωπίζει προβλήματα στην δουλειά του εξαιτία ε, του γεγονό ότι και οι δύο πλευρέ του αρνούνται πρόσβαση, που βάλουν περιορισμού, υπάρχουν ναρκοπαίδια κλπ. Ε, ταυτόχρονα, ε, υποστηρίζοντας ενώ υποστηρίζουμε τις διεθνείς προσπάθειες καλούμε την Ρωσία να επηρεάσει τους, ε, τις ομάδες των αποσχιστέντων ε, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι μισθοφόροι, ο στρατός και ο, στρατιωτικό στρατιωτικός εξοπλισμός από την Ανατολική Ουκρανία. Η, το πακέτο του Μίνσκ προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για αυτά. Επίσης θα συνεχίσουμε να ζητούμε και από τις δύο πλευρές του πολιτική ομάδα εργασία να συμφωνήσουν χωρίς καθυστερήσεις ε, τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν χώρα οι τοπικές εκλογές ε, στη, στο Ντονέτς και στο Λουγκάτς σύμφωνα με την Ουκρανική νομοθεσία ε, της προδιαφέρειας του ΟΑΣΕ ε, και με διεθνεί διεθνείς παρατηρητές. Ε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η πρόσβαση προφανώς ως βασικός όρος για να γίνουν εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις διεθνείς ε, προσπάθειες και είναι πρόθυμη να παίξει ε, ρόλο στην εφαρμογή των συμφωνίων του ΜΙΣΚ. Ε, η Αντιπρόεδρος κ. Μογκερίνη πρόσφατα ε, μετά την άτυπη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου των Υπουργών Εξωτερικών ε, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει περισσότερα συμπεριλαμβανομένη και τη στήριξη του πληθυσμού που επηρεάζεται άμεσα από τη σύγκρουση καθώς επίσης και τις μελλοντικέ εργασίες ανοικοδόμησης κατόπιν της εφαρμογής συμφωνίας του Μίνσκ. Επίσης είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και άλλα τμήματα της Συμφωνία του Μίνσκ. Για παράδειγμα, διενέργεια τοπικών εκλογών σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας όταν ε, πληρούνται οι όροι του ΟΣΕ. Ε, επίσης δίνουμε μεγάλη σημασία στην αστυνομική επιχείρηση του ΟΣΕ. η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι, τα κράτη-μέλη στηρίζουν την ε, ομάδα ε, παρακολούθησης του ΑΣΕΠΗ τόπου και θα αυξηθεί μάλιστα αυτή η στήριξη. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι μεγάλοι αριθμοί ατόμων που έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι προσιλωμένη στο να διατηρήσει στο ραντάρ της διεθνούς κοινότητας την ανθρωπιστική κρίση εκεί. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει χορηγήσει 66 εκατομμύρια ευρώ. Όμως περιορισμοί των ανθρωπιστικών ε, ενεργειών σε περιοχές που δεν έρχονται από την κυβέρνηση μας δημιουργούν ανησυχίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει σε όλα τα επίπεδα η ανθρωπιστική βοήθεια και σε αυτές τις προσπάθειες να δοθεί έτσι ώστε να είναι ένα πρώτο βήμα που θα οδηγήσει σε μια διαδικασία συμφιλίωσης. Η πρόσβαση και η κυκλοφορία των πολιτών από και προς τις μη ελεγχόμενες από τις κυβέρνηση περιοχές είναι επίσης ε, θέμα που μας δημιουργεί ανησυχίε. ανησυχίες. Ε, η ε, Ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει τις, τα κοινωνικά επιδόματα που είχαν ανασταλεί πέρσι. Στην τελευταία στις στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου έλαβε η χώρα στο Κίεβο ε, η συνεδρίαση ε, της Μικτής Επιτροπής Ουκρανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί επελέχθη μια ιδιαίτερα φιλόδοξη ε, διατύπωση για αυτό το θέμα. Παρόλο ότι δεν εστιαζόμαστε σε αυτό σήμερα. Ε, από πλευρά ασφάλεια, πρέπει να αναφερθούμε και στι εξελίξει στην Κρυμαία και τι ανησυχίε για την ασφάλεια εξαιτία της ε, αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της Κρυμαία τη Χερσονήσου. Η κυρία Μογκερίνη έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε αυτό το θέμα, συμπεριλαμβάνωμένη και της δήλωσης επί τη ευκαιρία της δεύτερης επαιτίου της ε, παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας που εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου. Ε, επίσης τον Αύγουστο όταν αυξήθηκαν οι εντάσεις ε, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μίλησε και στον Υπουργό κ. Κλίμκιν για αυτό το θέμα. Τέλος, δύο λέξεις για το διάλογο. Η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ θα συζητηθεί με την Ουκρανία στην Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανία που θα λάβει χώρα 24 Νοεμβρίου ε, στο Συμβούλιο Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανία στι 19 ε, Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Thank you, sir. Ευχαριστώ. Στο συντονιστές θα δώσουμε πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς έχω ένα ερώτημα για τις προβλέψεις σας για το άμεσο μέλλον. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις ε, ε, συνθήκες. Όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα κλιμακωθεί αυτή η ε, σύγκρουση. Σας η άποψή σας ποια είναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, εκτιμώ την απόφαση που πήρατε σε επίπεδο ΣΕΝΤΕ να ταξιδέψουμε στο Κίεβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, όσο πιο ανατολικά πάει κανείς από το Κίεβο, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα, αλλά καλό είναι να έχουμε μια άποψη επιτόπου και να έχουμε πληροφόρηση από αξιόπιστες πηγές. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάρτινς και θα ήθελα να τον ρωτήσω Γνωρίζετε τους λόγους γιατί υπάρχει τόση καθυστέρηση για τη συνάντηση στην Ορμανδία. Ε, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει τη θέληση, τη διάθεση να έρθει στο τραπέζι στα πλαίσια της συνάντησης της Νορμανδίας. Ίσως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν τους κατανοούμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το δεύτερο μου σημείο. Πώς αξιολογείται τον αντίκτυπο της έρευνας που ξεκίνησε το Μάρτιο, στις 17 Μαρτίου. Υπάρχουν κάποιες εκθέσεις ήδη, αναμένουμε και την ε, τελική. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν δημοσίως πριν από λίγες εβδομάδες. Εσείς πώς κρίνετε αυτή την κατάσταση υπό το φως και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και τι δράσεις ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει για να μπορέσει να αντικατοπτρίσει αναλογικά τα ευρήματα αυτά και να αναλάβει και, τη, και να προωθήσει και την ε, ε, αρχή της απόδοσης ευθυνών. αυτή που φταίνε θα πρέπει να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Σημαντική συμβολή σας. Θέλω και εγώ να πω κάτι και να συμπληρώσω ίσως λίγο και τις δύο παρεμβάσεις. υπήρξε μια πρόταση να πάμε όντω και πιο ανατολικά στην ε, Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Υπήρξαν προσπάθειες ε, και από τους προβλευτές ε, και από τη Γραμματεία. και του Προεδρείου τελικά του Κοινοβουλίου αποφάσισε να μην εγκρίνει αυτή την επίσκεψη. Για να είμαι ειλικρινής βέβαια, φοβούμαστε λίγο το... να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα γιατί μιλούμε για, τις... Ε, για τη διατήρηση των εκλογών. Αν θέλουμε οι Ουκρανοί να έχουν τη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να δούμε και την ε, σημασία, την αξία αυτής της επίσκεψης. Εμείς έχουμε την ασυλία μας, αλλά ακόμα ε, θυμάμαι το στρατιωτικό νόμο και πόσο δύσκολο ήταν στην ε, Πολωνία να έρθει κανείς σε επαφή με κοινοβουλευτικούς και να δει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι καταρχάς ασφαλής η επίσκεψή μας, δεν πάμε να εξερευνήσουμε, θέλουμε να δούμε τι περιορισμοί υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Και γνωρίζω ότι υπάρχει μια τάση οι αποστολές σε δύσκολες περιφέρειες, σε ζώνες μάχης. Είναι ίσως και λίγο θέμα ιδιωτικό, προσωπικό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε έγκριση και από τους υπολείπους για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε συνεπή ευρήματα. Και βεβαίως θα ήθελα, κύριε Μάρτινς, και εσείς να μας πείτε τι γίνεται με την ασφάλεια. Προφανώς είναι ε, πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς το οτιδήποτε, αλλά πείτε μας ε, εσείς ίσως για κάποια μέρη που θα ήταν ίσως καλό να πάμε. Ήδη έχουμε καταγράψει εμείς κάποιες περιοχές που ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικό κλίμα στις συζητήσεις, αλλά υπάρχουν διάφορες, ε, διάφορες ανησυχίες ό,τι αφορά την ασφάλεια των διαφόρων τμήματων, των διαφόρων σημείων, πόλεων της Ουκρανίας. Έχετε το λόγο. Ναι, να αρχίσω με, την, με τον αντίκτυπο της έρευνας της 17ης Μαρτίου. Ε, είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για τον αντίκτυπο αυτής της έρευνας, γιατί η έρευνα αυτή συνεχίζεται. Ήδη βεβαίω υπάρχουν κάποια ενδιάμεσα προσωρινά ευρήματα τα οποία έχουν δημοσιευθεί από αυτή την ποινική έρευνα. και ήδη μας βοηθούν να κατανοήσουμε ότι η έρευνα αυτή για την πτήση MH17 ε, δείχνει ότι το αεροπλάνο ε, καταρρίφθη από ρωσικό πύραυλο. στην ε, περιοχή των, που ελέγχεται από τους αυτονομιστές. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, ε, οποιαδήποτε υπόθεση πέραν αυτής της, αυτού του δεδομένου, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. θέλετε, τώρα μου είπατε συμβουλές για το ποιες είναι οι περιοχές που θα μπορούσατε να επισκεφθείτε. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή απάντηση, αλλά μπορώ να σας ε, στείλω την απάντηση, γιατί πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με την ε, αντιπροσωπεία μας επιτόπου, για να σας απαντήσω. Τώρα, για την ε, κλιμάκωση των συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Γερμανία και τη Γαλλία αναπτύσσουμε όλες τις δυνατότητες τις ε, διπλωματικές για να ε, αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακόμη και αν η σύγκρουση ε, συνεχιστεί είτε σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό για κάποιο καιρό, τώρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά βεβαίω θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την αποκλιμάκωσή τη. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, δεν έλαβα απάντηση για το πρώτο τμήμα της ερώτησής μου. Γιατί έχει αναβληθεί η συνάντηση στη Νορμανδία, γιατί αναβάλλεται κάθε φορά. Και επιπλέον, η αποστολή του ΟΑΣΕ ίσως δεν ήταν τόσο αποτελεσματική. Υπάρχει μήπως κάποια σκέψη να υπάρξει παράταση της α, ε, αποστολής της α, ε, CSDP. Γιατί ξέρετε, πρέπει να είμαστε αρκετά καινοτόμοι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τις ε, ε, εξέλιξει και να μην αφήσουμε πάλι να κλιμακωθεί η ένταση. Ευχαριστώ. Όντω έχει τεθεί αυτό το θέμα πολλές φορές γιατί ήταν και αίτημα τη Ουκρανική πλευράς η οποία παραπονεί το ακριβώς για τα ίδια πράγματα που μόλις αναφέρατε κι εσείς. Κύριε Μάρτινς, έχετε το λόγο για να απαντήσετε το πρώτο μισό της προηγούμενης ερώτησης. Οι λόγοι για την καθυστέρηση για τη συνάντηση της Νορμανδίας δεν είναι γνωστοί επισήμως. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, αν επισήμως, είναι ότι κάποια από τα μέρη θεωρούν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ε, επαρκής, για να υπάρξει επαρκής πρόοδος. Αλλά αυτό ατύπως το ξέρουμε επισήμως δεν γνωρίζουμε. Για το δεύτερο ερώτημά σας τώρα, για την ε, αποστολή CSDP. Ε, ναι. Είναι ε, ερώτημα που επαναλαμβάνεται και από την Ουκρανική πλευρά. Έχει αξιολογηθεί ήδη από την ΕΕΔ. Έχει συζητηθεί με τα κράτη-μέλη. Και το αποτέλεσμα είναι ότι προς το παρόν δεν θεωρείται η καλύτερη επιλογή. Η διεξαγωγή αυτή τη συνάντηση στην Ορμανδία. Το έθιξαν οι Ουκρανοί κατά τη διάρκεια της ε, συνάντησης PSC ε, στο Κιεβό. Νομίζετε, δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό. Μπορώ να θέσω εγώ παρακαλώ ένα ερώτημα ακόμη. Η τρέχουσα κατάσταση ασφάλειας, πώς πιστεύετε ότι επηρεάζει τα διάφορα προγράμματα τομεακά και μη που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία και τι πιστεύετε εσείς σχετικά. Πραγματικά επηρεάζει την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας Η δική μα υπηρεσία προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΚΟ, δίνει συνεχώ ειδήσει ότι έχει δυσκολία πρόσβαση σε περιοχές όπου δεν ελέγχει η κυβέρνηση. Ο αριθμός οργανώσεων που έχουν δικαίωμα να λειτουργούν είναι πολύ περιορισμένος και έχουν και πολλούς περιορισμούς στη λειτουργία τους. Αποκλείεται λόγω χάρη να εκδιπλωθεί οποιαδήποτε είδους βοήθεια με ευρωπαϊκή σημαία και ακόμη και με ευρωπαϊκή σημαία υπάρχουν περιορισμοί. Στις περιοχέ όπου υπάρχει έλεγχο τη κυβέρνηση δεν υπάρχουν ε, περιορισμοί. 1,2 δις ευρώ είναι η δική μας η πρόβλεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά τώρα έχουμε προβλέψει νέα ειδικά μέτρα για το 2017 120-200 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον μέχρι το τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών. Ε, μέχρι τώρα ε, στο παρελθόν είχαμε τις 200 εκατομμύρια, αλλά η επίσημη, εκταμίευση, το η επίσημη δέσμευση για την Ουκρανία είναι 120 και θα βρούμε τα υπόλοιπα κονδύλια ε, με άλλους τρόπους. Τι μέρος των προγραμμάτων αυτών θα ανασταλεί λόγω της ε, έλλειψης πρόσβασης. Έχετε κάνει υπολογισμού. Τα δύο τρίτα περίπου της ανθρωπιστικής βοήθειας παρέχονται σε περιοχές που δεν είναι υποκυβερνητικό έλεγχο. Δύο τρίτα από τα 66 εκατομμύρια που ανέφερα. Ε, αυτά εκταμιεύονται. Ε, τα εμπόδια και οι φραγμοί υπάρχουν αλλά ακόμα αυτό δεν έχει υπάρξει φραγμός, ε, ανάχωμα στη δράση μας. Ευχαριστούμε. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν μια πολύ μακρά ημέρα συζητήσεων, διαλόγου διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρτίν για την ε, παρουσία του εδώ και τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν μια ενημέρωση πρωτού πάει η Σέντε στο Κίεβο και ενδεχομένως στην Ανατολική Ουκρανία. Θα θέλαμε να έχουμε συναντήσεις με αξιωματούχους το ανώτερο επίπεδο, να είναι μια επίσημη επίσκεψη και να πάμε όλοι μαζί, όχι να κάνει ο καθένα ιδιωτικό τι επισκέψει του. Βεβαίω ενθαρρύνουμε και αυτού του είδου τι πρωτοβουλίε για τον κάθε βουλευτή. Είναι ε, δυνατόν, επιτρέπεται και είναι μέρο τη θητεία του τη αρμοδιότητα του κάθε βουλευτή. Όμως είναι πολύ δύσκολο μετά να καταρτήσουμε τις εκθέσεις μας και τα επίσημα έγγραφα για την επενημέρωση από τέτοιου ε, αποστολή. Δηλαδή, αυτέ οι ιδιωτικέ δραστηριότητες κάπου χάνονται στη σωρία των ε, δημόσιων γράφων που πρέπει να συνταχθούν μετά. Οπότε, καλό θα ήταν να έχουμε στο δυνατόν περισσότερη συμμετοχή στην επίσημη επίσκεψη της ΕΝΤΕ στην Ουκρανία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλου του ε, βουλευτέ και τους υπόλοιπους ε, προσκεκλημένους μας που ε, παρέστησαν και να έρθετε και αύριο. Έχουμε ακόμη σημαντικά σημεία να συζητήσουμε αύριο το πρωί. Ευχαριστώ.